δήλωση μάλλον της Επιτροπής Δυνάμει του άρθρου 231 σημείο 4 σας ενημερώνω ότι κατόπιν της τροποποίησης στις 5 το βράδυ εχθές